Η επόμενη συνεδρία στη Θελάβη χώρα αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 2 και το απόγευμα επίσης θα συνεχιστεί και τα πρακτικά είναι διαθέσιμα στην στοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συνεδρίασή μας.